δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Δίνω το λόγο στον κύριο εισηγητή για τέσσερα λεπτά. E, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν ε, στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής που συντάχθηκε κατόπιν δική μου πρωτοβουλία. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους κοιόδες εισηγητέ, ε, τι γραμματείες, ε, του συνεργάτε μα, ε, καθώ και τον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του εκπροσώπους και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Πάνω απ' όλα θέλω όμω να ευχαριστήσω τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και του εργαζομένου που μα στήριξαν σε πολύ μεγάλο βαθμό να αξιολογήσουμε αυτό το ταμείο. Τι είναι, είναι ένα ταμείο ένα ίδρυμα το οποίο ε, θεσπίστηκε ε, κατά το βελγικό δίκαιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη με τη συμμετοχή και άλλων ε, φορέων. Η Πολική Προεδρία είχε υποβάλει τη σχετική πρωτοβουλία, τη σχετική πρόταση το 2011 και τα δύο τελευταία χρόνια λειτουργεί αυτό το Ταμείο. Και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε ήταν διότι τα κλασικά εργαλεία για την υποστήριξη της δημοκρατίας είχαν αποτύχει, για παράδειγμα στη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης ή για την ε, ε, περίπτωση κάποιων ε, άλλων γεγονότων που είχαμε στα σύνορά μας προς Ανατολάς, Ανατολικά σύνορα. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στις στις ανατολικές χώρες και στις ε, κέντρο ευρωπαϊκές όπως την Πολωνία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο λοιπόν δημιουργήθηκε για να δρά ταχύτερα από τα προηγούμενα εργαλεία και να υποστηρίζει όσους δεν είχαν πάρει αυτή την υποστήριξη νωρίτερα. Και η δράση του είναι επιτόπου στις χώρες. Πάνω από 186 πρωτοβουλίες έχουν υποστηριχθεί σε όλες τις ε, χώρες ε, που βρίσκονται ε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από τους δικαιούχους θέλω να, ε, να τον αναφέρω είπε ότι μετά την Επανάσταση εγκαταλείφθηκαν όλοι, δεν λαμβάναμε πλέον χρήματα από πουθενά Ήρθε όμως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία με νοπά χρήματα και μας παρέχει όχι μόνο υποστήριξη αλλά και ιδέες. Αυτό λοιπόν είπε ένα ακτιβιστή από την Αίγυπτο συγκεκριμένα. Όσοι λοιπόν έχουν ε, πάρει υποστήριξη από αυτήν την ε, αρχή, από αυτό το ταμείο, παίρνουν και μέσω της ε, νομιμοποίησης, δηλαδή κάποιοι οποίοι υπονομεύονταν, στην Ουκρανία για παράδειγμα, και, και διώκονταν, είναι βουλευτές. Είναι βουλευτές σήμερα στο Βουλή της Ουκρανίας. Παρέχει λοιπόν μια μεταβατική χρηματοδότηση αυτό το ταμείο, γιατί χρηματοδότηση από το ένα παραδοσιακό ταμείο στο άλλο είναι χρονοβόρα διαδικασία και η προχρηματοδότηση επίσης ε, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Άρα με τον τρόπο αυτό ξεπερνάμε αυτά τα εμπόδια. Είχαμε διάφορα, διάφορες ε, συνεδριάσεις και ακροάσεις διοργανώθηκαν για να αξιολογήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Είδαμε και συνομιλήσαμε με δικαιούχους, ανταλλάξαμε εμπειρίες, δώσαμε και ε, ε στο προσωπικό του Ταμείου με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΕ. Τα δύο τελευταία χρόνια στην έκθεσή μας τα μελετήσαμε και διαπιστώσαμε ότι το Ταμείο πραγματικά ανταποκρίνεται στην εντολή του. Ιδίως την εντολή που του έχει ε, αναθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και συνιστά πραγματικά ε, προσθέμενη αξία σε αυτή την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, προαγωγή της δημοκρατίας ανά τον κόσμο το Ταμείο θα πρέπει να τύχει της ε, κατάλληλης ε, οικονομικής στήριξης ε, και χαιρετίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρία χρόνια προβλέπεται πλέον να λάβει χρηματοδότηση αυτό το Ταμείο. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ξεκινάμε τη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑ. Ήθελα να δώσω το λόγο σε όλου, αλλά σα παρακαλώ να διατηρήσετε το χρόνο. Ο κύριος Πόσπιτζελ έχει το λόγο και επειδή δεν μπορούσα να τον δώσω προηγουμένω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον συντάκτη της έκθεσης. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υποστηρίξει τις ΜΚΑΟ σε χώρες ε, που υφίστανται πολιτικές μεταβολές. Εγώ είμαι βουλευτής της Τσεχικής Δημοκρατίας, η οποία έχει κομμουνιστικό παρελθόν και εγώ υπήρξα μέλος πολλών τέτοιων οργανώσεων. Χωρίς τα χρήματα από Ιδρύματα της Δυτικής Ευρώπης δεν θα είχαμε καταφέρει να διοργανώνουμε διασκέψεις και εκδηλώσεις και δεν θα είχαμε καταφέρει να, φέρουμε, ε, να ενημερώνουμε τον κόσμο στην Τσεχική Δημοκρατία. Είναι σημαντικό αυτό, δεν αποτελεί απλά ένα διανομή χρήματο. Είναι ηθική μα υποχρέωση, ειδικότερα στι χώρε τη ε, πρώην ε, Σοβιετική Ένωση και στη Μέση Ανατολή, όπου δεν υπάρχει στη βαρύ δημοκρατία. Ελπίζω οι 12 χώρε που δεν έχουν ακόμα πληρώσει τη συμμετοχή του να το πράξουν μετά από τη σημερινή έκθεση, γιατί όπω είπα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία έδειξε μετά από δύο χρόνια ύπαρξης ότι έχει εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες, την ελευθερία, τη δημοκρατία και έχει πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα. Το EED παραμένει ένα ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου που παρέχει ευέλικτα αποτελέσματα, ευέλικτη χρηματοδότηση βάσει της ζήτησης απευθείας τους δικαιούχους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο που συμπληρώνει και τα άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελάχιστο διοικητικό φόρτο και απλές διαδικασίες. Είναι ζωτική σημασία για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του ΙΕΔ, να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη, σταθερή, προβλέψιμη και διαφανή χρηματοδότηση. Θα ήθελα να κάνω έκκληση για τις ομάδες ε, ε μας να υποστήριξουμε όλες τις ομάδες ε, μειονοτήτων, LGTB, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να τους στηρίξει όλους αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεμέσμακερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Ξύπ για την έκθεσή του και ε, εγώ είμαι μαζί του στο ε, ε, Διοικητικό Συμβούλιο και χαίρομαι που είναι ένα ταμείο που δραστηριοποιείται στη γειτονία. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία των πολιτών. Στην Ουκρανία έχει μικρούς εταίρους που ε, έλεγαν και τους υποστήριζε που έδιναν ειδήσει από το Euromaidan στο Κίεβο. Υποστηρίζει bloggers, δημοσιογράφους, ακτιβιστές στο Αρμπαϊτζάν, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο που ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης υφίσταται ακόμα μεγάλη πίεση. Στις χώρες γειτονίας και αλλού η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα υφίσταται ένα πόλεμο προπαγάνδας που ε, εκπορεύεται από το Κρεμλίνο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο μπορεί να μας βοηθήσει. Γιάκοφσιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ε, το ταμείο αυτό δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Διότι είχα και εγώ προσωπικά την ευκαιρία να ε, συμμετάσχω σε διάφορες ε, προσπάθειες σε σύσταση διαφόρων ιδρυμάτων και είδα τι αποτελεσματικότητα έχουν και πόσο τόπο πιάνει η δουλειά τους σε γειτονικές μας χώρες. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε τις υποψήφιες χώρες ή τις δυνάμει υποψήφιες χώρες. Και εδώ αναφέρομαι εγώ κυρίως χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τις οποίες γνωρίζω καλύτερα. Γνωρίζω την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές και την κατάσταση που επικρατεί στα μίντια. Έχουν υποχρηματοδότηση, έχουν προβλήματα, ιδιαίτερα μικρά, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Ε, είναι τεράστια λοιπόν η βοήθεια που δέχονται από το Ταμείο ε, για να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και να μην υποκύπτουν σε πιέσεις. Ο κύριος Μπουτικόφερ. I Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ε, ευχαριστώ σε τρεις πλευρές. Πρώτον, ευχαριστώ τους ε, δημιουργούς αυτής, τους εμπνευστέ αυτής της πρότασης, τους Πολωνούς. Δεύτερον, ευχαριστώ όσους έχουν εργαστεί με το Ταμείο για να καταστεί επιχειρησιακό. Και τρίτον, και εξίσου σημαντικό, ευχαριστώ κύριε Γκριτζίμπ, κύριε Σιγητά, που συνεργαστήκατε με όλους και όλες εμάς για να καταθέσετε μια αρτιότατη και πολύ θετική έκθεση. Το ευέλικτο μέσο το οποίο παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο τη Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις όπου περισσότερες συνεχώς χώρες δυσκολεύουν τις οργανώσεις τον των πολιτών όλο και περισσότερο όπως και τις μη ε, ε, κυβερνητικές οργανώσεις να διδραματίσουν έναν δημοκρατικό ρόλο όπως θα έπρεπε στις ε, κοινωνίες των χωρών τους. Εμείς μέσω του Ταμείου μπορούμε να προστατεύσουμε τις οργανώσεις αυτές και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προαγωγή της δημοκρατικής Και τελευταία πρόταση. Προσθέτω και εγώ τη δική μου φωνή σε όσους ζητούν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοθούν. Διακόπτεται. Ο επόμενος ομιλητής είναι Κορεάο. Κορεάο, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ε, ε, σκιώδης συζητητής ε, ήδη συζήτησα με τους συναδέλφους για την ποιότητα αυτού του κειμένου, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι για το οποίο θα πρέπει να πιστήσουμε την προσοχή αυτή τη στιγμή επειδή ο, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζονται οι χρηματοδοτήσεις αυτές ε, γίνεται σε ένα γραφείο της Προεδρίας ε, το οποίο σύνθεση δεν αντιστοιχεί στις δυνάμεις αυτού του Κοινοβουλίου. Εμείς ζητήσαμε λοιπόν με μια τροπολογία το board ε, που λαμβάνει αποφάσεις για τα χρηματοδοτήσεις αυτές να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η γκουε, e, δεν υπάρχει το EFTD και δεν υπάρχει και η νέα ομάδα. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να διδάσκουμε τη δημοκρατία πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε δημοκρατικά τη σύνθεση του Κοινοβουλίου διότι αλλιώς ε, ε, κάνουμε πλάκα. Ε, θα πρέπει να υποστηρίξετε αυτή την τροπολογία στην οποία βασίζεται η εξοπιστία του Ταμείου αυτού το οποίο αποτελεί το αντικείμενο επίκριση από εμά. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Κίνκαγκάλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κρίσ για την εξαιρετική του δουλειά για το EED. Όπως φαίνεται δημιουργήσαμε ένα εργαλείο ευέλικτο, προσαρμόσιμο σε επίγουσες καταστάσεις και σε νέες καταστάσεις και αποτελεσματικό. Χαίρομαι που από δική πρωτοβουλία έχουμε τις εθνικές και γλωσσικές μειονότητες ε, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τις μειονότητες στην Ουκρανία για παράδειγμα ώστε οι κοινότητες τους να ε, ε, ενδυναμωθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επίσης σημαντικό είναι δεδομένο των πρόσφατων γεγονότων η ελευθερία των θρησκευτικών πεπιθήσεων να αποτελεί επίσης να λαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για να προστατεύσουμε τις μεγάλες ομάδες χριστιανών που αποτελούν θύματα επίθεσης. Ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε τρία θέματα θέλω να θίξω. πρώτα απ' όλα η ίδρυση του ευρωπαϊκού ταμείου για τη δημοκρατία είναι μια σημαντική δραστηριότητα διότι μπορεί μέσα από τις δράσεις του ταμείου να υπάρξει στήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλων δράσεων. όμως δεύτερη παρατήρηση δεν θα πρέπει το ταμείο αυτό να αξιοποιείται ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και επέμβασης στα εσωτερικά άλλων κρατών γιατί αυτό θα οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα. και το τρίτο μου κάνει εντύπωση έγιναν 186 δράσεις από το ταμείο αυτό. Καμία από τις δράσεις αυτές δεν ασχολήθηκε με τη στιγμή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες του Μνημονίου. Έχουμε ειδική έκθεση του Κοινοβουλίου μας το Μάρτιο του 2013 που λέει ότι η Τρόικα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Δεν είδα μία δραστηριότητα του Ταμείου αυτού ας αποκαταστήσουμε τη λειτουργία των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ένωση και ευχαρίστως βεβαίως να ασχοληθούμε και με θέματα αντίστοιχα σε άλλες χώρες. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία Κατσέα και θέλω να δώσω το λόγο στην Επίτροπο την κυρία Μάνσον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με μεγάλη χαρά εξ ονόματος ε, της κυρίας Μογκερίνη λαμβάνω το λόγο εδώ για να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους υπολείπους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ για τη σημαντική σας εργασία στην αξιολόγηση του έργου του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ευρεία υποστήριξη του έργου αυτού ε, ανεξαρτήτως πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου και είναι σημαντική η δική σας εργασία στο Διοικητικό Συμβούλιο και τρόπος με τον οποίο διαδραματίζεται πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση και στη διάδοση του έργου του. Συμφωνώ με την έκθεση ότι το Ταμείο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό γιατί υποστηρίζει τη δημοκρατία στη γειτονιά μας και είναι χρήσιμο εργαλείο που έχει ε, να, έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της. Όπως λέτε και εσείς, ε, δίνει υποστήριξη ταχεία όσο και ευέλικτη ε, σε επιθετικό περιβάλλον όπου πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να φτάσει στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δίνει ε, επίγουσα βοήθεια ε, και το Ταμείο να υποστηρίζει ε, μικρούς δικαιούχους που δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεγαλύτερα προγράμματα. Είναι λοιπόν συμπρωματικός ο ρόλος του, θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο το Ταμείο και να έχει το περιθώριο εκείνο που χρειάζεται για τις κινήσεις και το έργο του. Στην έκθεσή σας κάνετε προτάσεις για την αναθεώρηση και σας διαβεβαιώ ότι συμμετέχει και το Ταμείο στην αναθεώρηση της ε, πολιτικής γειτονίας και είχε την ευκαιρία να κάνει προτάσεις και συστάσεις πολύ συγκεκριμένες όσο και χρήσιμες και μάλιστα αυτό βασίζεται ε, στις απόψεις των δικαιούχων. Η κοινωνία των πολιτών στη γειτονία μας ε, έχει ακολουθήσει τη συζήτηση και μπορεί να την τροφοδοτεί κιόλα. Είναι θετικά τα αποτελέσματα λοιπόν της ε, αξιολόγησης του Ταμείου όπως και η σύστασή σας προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι στην υποστήριξη αυτή του έργου. Θα ήθελα να σας πω ότι μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε περαιτέρω 12 εκατομμύρια χρηματοδότηση για την επόμενη διετία 2016-2017 και αυτή είναι σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρηματοδότηση. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι έχει σημασία το Ταμείο αυτό να ε, συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέσα και εργαλεία και να ε, χρηματοδοτεί δικαιούχους που δεν ε, είναι επιλέξιμοι για τα λοιπά ταμεία. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και ε, δίνει βοήθεια με βάση τη ζήτηση. Θα συνεχίζουμε να το διαφημίζουμε το προσωπικό μας και να συνεχίσει το καλό του έργο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή και προσβλέπουμε στη συνέχεια της καλής μας συνεργασίας επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, ε, για τα καταληκτικά λόγια και συγχαίρω τον κύριο Ξύπ για την έκθεσή του. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνω τη συζήτηση. Ακολουθούν οι ψηφοφορίες αμέσως μετά στις 12 η ώρα ακριβώς. Λίγα λεπτά μέχρι τις 12. Καλώς διαχειριστήκαμε το χρόνο. Μικρή λοιπόν διακοπή της συνεδρίασης. Ja. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Ερχόμαστε στις ψηφοφορίες, παρακαλώ καθίστε. για να προλάβω να μην ζητάτε το λόγο. Είναι πάρα πολλές οι ψηφοφορίες και χρειάζεται να ψηφίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση και προσήλωση. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, η διάρκεια των ψηφοφοριών έχει επιμηκυνθεί διότι ζητήθηκαν πάρα πολλές ψηφοφορίες κατά τμήματα και χωριστές. Κυρία Άουκεν. Ε, ε, Ο πρόεδρος Σούλτς μας υποσχέθηκε χθες ότι θα είχαμε ενός λεπτού σιγή για τους ε, όσους σκοτώθηκαν πέρυσι στη Γάζα χιλιάδες παιδιά. Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε τώρα. Ο Σούλτς είπε σαφώς χθες ότι θα διατηρούσαμε ενός λεπτού σιγή και το συζητήσαμε χθε το βράδυ μάλιστα μαζί του. Κυρία Όκεν, ο πρόεδρος είπε και το τσέκαρα ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται έτσι άρον-άρον. Θα πρέπει να το προετοιμάσουμε σωστά και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση ποιετικά είναι. Κυρία συνάδελφε. I Πώς ελήφθη αυτή η απόφαση. Εχθές ελήφθη απόφαση για ενός λεπτού σιγήν ε, επιτόπου την ώρα που το ρωτήσαμε. Η καινούργια απόφαση πώς προκύπτει. Μα αν με είχατε ακούσει θα ξέρατε για ποιο λόγο. Μπορείτε να με ρωτήσετε διμερώς στη συνέχεια και θα σας εξηγήσω. Δεν πρόκειται να λάβω τώρα κανέναν άλλο συνάδελφο. Όποιο θέλει να μιλήσει για αυτό το θέμα θα το διακόπτω. Κύριε Βούλφ. This is just a, a procedural issue. Ένα διαδικαστικό ζήτημα μετά από τις εξηγήσεις ψήφων χθε. Θα μπορούσε να μας εξηγήσει ο Πρόεδρος τι θα συμβεί μετά από αυτή τη συζήτηση με τις χθεσινές αιτιολογήσεις ψήφου και τις σημερινές. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Μετά τις ψηφοφορίες θα ακούσουμε τις χτεσινές πρώτα επεξηγήσεις και θα συνεχίσουμε με τις σημερινές και βλέπουμε. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Έκθεση. Ορίστε κύριε Ρούμπιχ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα μόνο να ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι οι ψηφοφορίες σήμερα θα διαρκέσουν πάνω από δύο ώρες. Είναι δυνατόν μήπως να αναβάλουμε καμία ψηφοφορία για μετά το καλοκαίρι. Δύο ώρες ψηφοφορία σήμερα είναι αυτά πράγματα. Κύριε Ρούμπιχ, δεν άκουσα εγώ για δύο ώρες. Μια μισή ώρα έχω προβλέψει. Γιατί εκεί δεν λαμβάνεται υπόψη ότι Ήδη χάσαμε τέσσερα λεπτά. Λοιπόν, πάμε. Έκθεση ποιοτικά είναι. Παράγραφο 1 σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτον ψήφι π. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Το αρχικό κείμενο τμήμα 1, Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.